της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να ζητήσω λοιπόν από την κυρία Υφυπουργό να λάβει και πάλι το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρώτα Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη, Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεμελιώνεται σε αξίες όπως ε, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτές είναι οι κοινέ αξίες των κρατών μελών και αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της ε, ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εσωτερική τάξη σέβεται πλήρως το κράτος δικαίου και άλλες θεμελιώδεις αξίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη αυτών των ουσιαστικών αρχών. Αναγνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πληρούν τα καθήκοντά τους. Όπως θα θυμάστε, τον Ιούνιο του 2013 το Συμβούλιο δήλωσε ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη συζήτηση βάσει των συνθήκων για την πιθανή ανάγκη και διαμόρφωση μιας ε, μεθόδου ε, συστηματικής ε, και μέσω συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Τους επόμενους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να τηρήσουν τις υποχρεώσεις της συνθήκης για τις θεμελιώδεις αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισέφερε σε αυτή τη συζήτηση με την ανακοίνηση το Μάρτιο του 2014 για το θέμα. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνουν ε, τα υφιστάμενα μέσα. Διαδικασίες επί παραβάση, οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβίασης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και ε, η δυνατότητα της ατομικής βόμβας που προβλέπεται από το άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία επιτρέπει την ε, αναστολή του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών και συνεχών παραβιάσεων των ε, ευρωπαϊκών αξιών. Το Συμβούλιο σε αρκετές περιπτώσεις συζήτησε πώς μπορεί να διαφυλάξει καλύτερα το κράτος δικαίου στην Ένωση. Το Δεκέμβριο πέρσι το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα τα οποία καθορίζουν έναν ετήσιο πολιτικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση και διαφύλεξη του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάλογος θα σέβεται κάποιες αρχές, όπως για παράδειγμα η αντικειμενικότητα, η έλλειψη διακρίσεων και η ίση μεταχείριση. Επίσης, θα σέβεται την αρχή της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα ακολουθείται μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τους πάντες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Προεδρία θα διαδραματίσει σημαντικό, ε, κεντρικό ρόλο για να διασφαλίσει ότι αυτές οι αρχές γίνονται σεβαστές σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο προετοιμάζει την πρώτη πολιτική συζήτηση για το θέμα του κράτους δικαίου ε, ε, στα πλαίσια του έτους. Είμαι πεπισμένη ότι ο διάλογος αυτός θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι το κράτος δικαίου θα συνεχίσει να αποτελεί μια κοινή θεμελιώδη αξία η οποία ε, καθορίζει την ένωση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε μια πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φραν Τίμεμαντ από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο σαφέστερο τρόπο να δείξουμε τι σημαίνει για μα το κράτο δικαίου στην καθημερινή ζωή είναι να θυμηθούμε τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει κράτο δικαίου. Όταν ο πρόεδρο Άιζενχάουερ σημείωσε την πρώτη τέτοια ε, εορταστική ε, επέτειο είχαμε ακόμη τι εικόνε και το φόβο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο μυαλό μας. Τώρα έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε και την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε το Γενάρη ακριβώς ε, ε, θυμηθήκαμε την απελευθέρωση των στρατοπέδων ε, συγκέντρωσης και πήγα και εγώ και ο πρόεδρος Σούλς στο Τερέζιεν Κάμπ αλλά αυτά που διαπιστώνουμε και τώρα αυτό το πλαίσιο προβλημάτων είναι μια έκκληση για επαγρύπνηση. επαγρύπνηση. Γι' αυτό καλωσορίζω αυτήν την συζήτηση. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να επαγρυπνούμε για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στις κοινωνίες μας ε, αργά και ανεπέστα να επανέλθουν σε ανελεύθερες λογικές. Δεν υπάρχει ανελεύθερη δημοκρατία. Η ένωσή μας βασίζεται σε μια σαφή ρήξη με το παρελθόν βασίζεται στην αρχή ότι οι κοινωνίες πρέπει να είναι ελεύθερες, να μην υπάρχει αυθαιρεσία των ισχυρών. Αυτό το μεγάλο βήμα είναι η βάση της Ευρώπης. Πολύ συχνά όλα αυτά τα θεωρούμε δεδομένα. Άρα πρέπει να επαναλάβω επανειλημμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη αν δεν υπάρχει πλήρη σεβασμό των ε, βασικών μα και κοινών μα αξιών, επί των οποίων δεν μπορεί να υπάρξει κανένα συμβασμό, γιατί θα είναι συμβασμό επί του ίδιου του ιστού τη ευρωπαϊκή συνεργασία, επί τη ίδια τη φύση Τη Ευρωπαϊκή Διαδικασία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Ο πρώτο Γιούνκερ ε, με εμπιστεύθηκε αυτά τα καθήκοντα. Τα καθήκοντα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Να συντονίσω την εργασία προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια εργασία καθημερινή. Η συμπερίληψη σε όλα τα θέματα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συστατικό στοιχείο τη νομοθεσία από την διατύπωσή τη μέχρι την έγκριση τη όπω ε, ε, συνολικά με, τον, με την Επιτροπή εγώ και ο κύριος Αβραμόπουλος είμαστε οι βασικοί αρμόδιοι για τα θέματα αυτά αλλά καλούμε και τους άλλους ε, επιτρόπους να συμμετάσχουν σε αυτή την εργασία αν χρειάζεται. Θέλουμε να εφαρμόζονται παντού και να προστατεύονται παντού σε όλα τα κράτη-μέλη τα θεμελιώδη δικαιώματα με βάση την προφόρηση που συλλέγουμε από κάθε κράτος μέλος επιτόπου. Ξέρουμε ότι το σώμα σας επανειλημμένα έχει καλέσει για να υπάρχει αποτελεσματική και δεσμευτική νομοθεσία που να συμπληρώνει το άρθρο 7 Όλοι συμφωνούμε επί των στόχων που είναι πίσω από αυτές τις εκκλήσεις. Θέλουμε οι κοινέ μας ε, αξίες να γίνονται πλήρως σεβαστές. Το βασικό θέμα είναι ποιος είναι ο καλύτερος στόχος για να επιτύχουμε, ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Για μένα όλα τα θεσμικά όργανα έχουν συμπληρωματικού ρόλου προ αυτή την κατεύθυνση. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένα ετήσιο διάλογο για το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι η συζήτησή μα σήμερα εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ίδιο στόχο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το ρόλο τη. Σύμφωνα με τι συνθήκε, τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει αποφασιστική δράση και έχει ασκήσει πολιτική πίεση και επιτυχημένα έχει απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περιπτώσει απειλών για τα βασικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, για την παράνομη συνταξιοδότηση δικαστών ή για μέτρα που θίγουν την ανεξαρτησία ρυθμιστικών αρχών και αρχών εποπτείας και κυρίως η νομοθεσία μας ασχολείται με θέματα συμβατότητας ε, κάποιων ε, θεμάτων ισχύω ε, του κράτους δικαίου. Για παράδειγμα, δυνατότητες προσφυγής υπάρχουν. Και τι πρέπει να γίνει αν ορισμένες αρχές δεν έχουν επαρκείς αρμοδιότητες ή ανεξαρτησία. Από τον προηγούμενο Δεκέμβριο υπάρχουν περισσότερα μέτρα στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας και για αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να εξετάσει εάν σέβονται τη θεμελιώδη ελευθερία. Θα κάνω ό,τι μπορώ τους, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με μη δογματικό τρόπο και να αποτιμά αντικειμενικά και αμερόληπτα κάθε περίπτωση ανάλογα με το γράμμα και το πνεύμα του, ρόλου, πρέπει, του νόμου. Πρέπει να δράσουμε αμερόληπτα και να αντιμετωπίσουμε ισότιμα όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανένα κράτος μέλος περσέ, αλλά να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα με βάση στοχευμένα μέτρα για να υπάρξει σωστή εφαρμογή του ενωσιακού νόμου. Το άρθρο 7 μας δίνει δυνατότητα να επιβάλλουμε ευρείες κυρώσεις. Δεν περιορίζεται σε τομείς που καλύπτει μόνο η ενωσιακή νομοθεσία. Είναι διατυπωμένο έτσι ούτως ώστε να αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όμως η εμπειρία μας από το παρελθόν μας έχει καταδείξει ότι αυτό το μέσο που μπορεί να πυροδοτηθεί από την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το 1 τρίτο των κρατών μελών, δεν είναι πάντα το καλύτερο για ταχεία αντίδραση. Υπάρχουν καταστάσεις που δεν είναι εντός του πεδίου εφαρμογή του νοσιακού δικαίου και δεν ικανοποιούν το κατόφλιο του άρθρου 7, αλλά μας ανησυχούν όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο, τον προηγούμενο Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτό το πλαίσιο κράτους δικαίου που καθορίζει πώς αντιδρά η Επιτροπή σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο με το κράτος μέλος αν διαπιστώνουμε συστηματικούς κινδύνους για το κράτος δικαίου για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Εάν υπάρξει μια τέτοια κρίση για το κράτος δικαίου, το πλαίσιο επιτρέπει στην Επιτροπή να αντιδράσει και ταχαίως, μετά από αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης και με πλήρη σεβασμό τη αρχή της ισότιμη αντιμετώπιση των κρατών μελών. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε λύση με το κράτος μέλος το συγκεκριμένα για να μην χρειαστεί να τεθούν σε ισχύ οι μηχανισμοί του άρθρου 7. Το Κοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό πολιτικό ρόλο για να στηρίξει τις προσπάθειες Επιτροπής να πείσει το κράτος μέλος να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή κράτου δικαίου. Το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά για τι πρόοδος έχει σημειωθεί σε κάθε φάση τη διαδικασία κάθε περίπτωση. Παρακολουθούμε από κοντά όλα τα παρόμοια θέματα που προκύπτουν στα κράτη-μέλη και δεν θα διστάσω να αξιοποιήσω το πλαίσιο αυτό εάν απαιτείται από την κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο κράτο-μέλο. Επευκαιρία να ασχοληθώ και με ένα συναφέ θέμα. Πολλοί από εσά μπορεί να διαρωτώνται τι γίνεται για την ε, ένταξη της Ένωσης στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι στόχος πάντα της Επιτροπής και μου προσωπικά αυτή η ένταξη. Νομίζω ότι θα ενδυνάμωνε τις κοινέ μας αξίες. Όμως η γνώμη του δικαστηρίου, η απόφαση του δικαστηρίου θέτει σημαντικές προκλήσεις. Ορισμένε δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια περίοδο εξέταση του προβλήματο, να κάνουμε τι διαβουλεύσει με όλου του εμπλεκόμενου για να δούμε ποια είναι η καλύτερη διέξοδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσόρισε το πλαίσιο αυτό και τις αιτήσεις συζητήσεις στο Συμβούλιο γνωρίζω ότι υπάρχουν νέες εκκλήσεις να υπάρξουν νέοι επιπλέον μηχανισμοί για την μόνιμη επιτήρηση του κατά πόσο συμμορφούνται τα κράτη-μέλη με τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαι πεπισμένο και η πρακτική μου ήταν πάντα ότι αν δεν επαρκούν τα υπάρχοντα μέσα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Και πάντα μπορώ να σκεφτώ πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το σεβασμό των αξιών μας. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε σε μακροχρόνιες συζητήσεις για ενδεχόμενα νέα μέσα και εργαλεία, πρέπει να δούμε τι διακυβεύεται. Μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας ότι χρειαζόμαστε και έναν επιπλέον μηχανισμό επιτήρησης κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού ή πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Η πείρα έχει δείξει ότι δεν χρειαζόμαστε νέους μηχανισμούς ή νέες εκθέσεις αλλά πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα της Ένωσης να δρά και να παρεμβαίνει σε ορισμένα είδη κρίσεων και περιπτώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, το πλαίσιο διαρθρώνεται με βάση τα κύρια θέματα. Και πολλά ε, προβλέπονται ήδη για ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων για τη συμμόρφωση στα κράτη-μέλη. Πολλοί συμπεριλαμβανομένων των θεσμών της Ένωσης και των οργανισμών της Ένωσης και ιδιαίτερα τον οργανισμό, του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που εργάζεται θαυμάσια πρέπει να πω, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Επιτροπή της Βενετίας και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι παρακολουθούν και αποτιμούν την κατάσταση. Η πληροφόρηση αυτή βέβαια πρέπει να είναι πιο προσβάσιμη. Και γι' αυτό στοχεύω για το ετήσιο σεμινάριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάτι που είπα κατά την ακρόασή μου. Στοχεύω λοιπόν αυτό το ετήσιο σεμινάριο να γίνει τον ερχόμενο Οκτώβριο, ίσω αρχές Νοεμβρίου. Και θέλω όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου, να συμμετάσχουν. Και θέλω να αναγγείλω εδώ, ενώπιόν σα ότι ω θέμα για το φετινό ε, σεμινάριο θέλω να προτείνω την αποδοχή των άλλων. Πώς να αντιμετωπίσουμε τις απόψεις που είναι κατά των μειονοτήτων, κατά των ε, χριστιανών, κατά των ε, Εβραίων, κατά των μουσουλμάνων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας σήμερα. Ελπίζω να βοηθήσετε σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση. Θέλω να γίνει ουσιώδη συζήτηση. Εάν μιλήσουμε από κοινού και αν διακηρύξουμε τις απόψεις μας από κοινού, στέλνουμε ισχυρό πολιτικό μήνυμα και πιστεύω ότι αυτό θα σήμαινε περισσότερο, περισσότερα για τους πολίτες μας από μακρές ενδο θεσμικές συζητήσεις. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ε, σύγκληση της κοινωνίας μας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον φόβο του άλλου, τον φόβο που μας παραλύει. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε την έννοια των κοινών μας αξιών. Δείχνουμε έτσι τι οφείλουμε στην ιστορία μας και τι θέλουμε να επιτύχουμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτή είναι η συζήτηση. Αυτά αναμένουν οι πολίτες μας από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε και εμείς ε, πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση. Ο κύριος Μπούντα λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Ζακ Σεβαλιέ ορίζει το κράτος δικαίως εξή. Πρόκειται για ένα πολιτικό σύστημα όπου η εξουσία του κράτους ελέγχεται από το δίκαιο. Το κράτος δικαίου ήταν και θα εξακολουθεί να είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση σε κάθε σύγχρονη κοινωνία. Αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ασφάλεια, τέτοιου είδου αξίες πρέπει να αποτελούν τον κοινό παρονομαστή σε μια ενωμένη και ασφαλή Ευρώπη να είμαστε όλοι στην υπηρεσία των ε, πολιτών και αυτές λοιπόν οι αξίες και στο μέλλον θα παραμείνουν αναπαλωτρίωτες. Μια σταθερή Ευρώπη με σταθερά κράτη αυτό σημαίνει ε, ασφάλεια για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την πρόλευσή τους. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αποτελεσματική δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις και για τις θέσεις απασχόλησης. Οποιαδήποτε απομάκρυνση από αυτές τις αξίες οδηγεί σε ανασφάλεια και αυτό επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί που οποτεδήποτε διαπιστώνεται παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών ε, θα υπάρχει και μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Οι αξίες ε, του κράτους δικαίου μπορούν πολύ εύκολα να αμφισβητηθούν και σε δημοκρατίες οι οποίες ε, θεωρούνται σταθερές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα αλλά και η Ρουμανία ειδικότερα κατέδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν τέτοιου είδους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ε, ασφάλεια του κράτους δικαίου. Ε, ένας ελεγκτικός μηχανισμός ε, επιτρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις κατά της ευνομίας. Εξάλλου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, τα κρατημέλη, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σωστές στρατηγικές στον τομέα της δικαιοσύνης. Και αυτά τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μία μπλε κάρτα, την δέχεστε από τον κύριο Σόνι. Παρακαλώ κύριε Σόνι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο αυτά που αναφέρατε. Και νομίζω ότι έπαιξε και ο κύριος Τίμερμανς, αλλά αγαπητέ συνάδελφε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής στο ΕΛΚ. Τα λέτε αυτά και στο Ογκουρικό κόμμα που ανήκει στο ΕΛΚ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο συνεχίζει να μιλάει. Μιλάει μονίμως για την ανελεύθερη δημοκρατία και επιβάλλει και διακρίση. Πρόεδρε, προφανώς και υπάρχει αυτή η συζήτηση σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Και κάθε χώρα θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες και σε επίπεδο συμβουλίου δεν θα πρέπει να υπάρχουν παραβιάσεις δημοκρατίας γιατί αυτό ε, συνεπάγεται κυρώσεις. Η κυρία Ζίπελ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το ευνομούμενο κράτος και η δημοκρατία είναι τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όποιος ταρακουνάει τα θεμέλια αυτά, ταρακουνάει κατ' ουσίαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σεβασμός των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων είναι νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών και αυτό όχι μόνο όταν εφαρμόζουν το ε, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντα. Πολύ συχνά όμως ε, ε, περιφρονούνται, υπάρχει περιφρόνηση έναντι αυτών των δικαιωμάτων, ισχύει για τη δικαιοσύνη και για τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διωγμοί αλλά και αποκλεισμοί των μειονοτήτων. Εμείς ως Ευρωπαίοι λοιπόν δεν μπορούμε απλά να παραμένουμε αδρανείς διαπιστώνοντας ότι περιφρονούνται θεμελιώδη δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συστήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για την παρακολούθηση εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη, απόλυτα ανεξάρτητη επιτροπή από οποιαδήποτε επιρροή. Μέχρι τώρα ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο κατέθεσαν επιστικά προγράμματα. Έχουμε τα ε, θέματα που συζητάνε τα κράτη-μέλη ε, όταν συναντιούνται σε μεσημεριανά γεύματα, θέματα που άπτονται των θεμελιδών δικαιωμάτων, ε, όμως αυτά πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης και το πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν για την προστασία του κράτους δικαίου, αυτά μέχρι τώρα παραμένουν κενό γράμμα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτάχων χρονικά διαστήματα για τα μέτρα που λαμβάνονται. Αυτό δεν έχει συμβεί είτε γιατί δεν ελήφθηκα ένα μέτρο, είτε γιατί δεν ενημερώθηκε το Κοινοβούλιο. Και συνοψίζω, μετά από τις συζητήσεις των τελευταίων ετών ε, για τα ε, δικαιώματα, τώρα το Συμβούλιο και Κομισιόν προσεγγίζουν, πλησιάζουν τις απόψεις τους. Ε, καλό είναι αυτό, αλλά δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε τη βούληση όλων των κρατών μελών να ονοματίζουν τις ε, παραβιάσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις. Νομίζω αυτή είναι η ευθύνη μας, ε, μια, η ευθύνη μιας ένωσης αξιών. Ευχαριστώ, ο κύριος Κύρκοπ, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, οι κοινέ αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοχής είναι φυσικά τα θεμέλια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει με επιστημονικό τρόπο αξίες οι οποίες δεν ποσοτικοποιούνται από την πείρα μου στη ζωή, οι πίνακες βαθμολόγησης, οι δείκτες, τα benchmarks, πολύ συχνά ελάχιστα αντανακλούν ε, την πραγματικότητα μιας ε, κατάστασης ή την ε, χαλαρώνουν το να χρησιμοποιούμε μέσα για να τιμωρούμε τα κράτη-μέλη και να παρέχουμε εργαλεία για πολιτικές βαθμολογίες ε, είναι κάτι το οποίο αντί αυτού θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε κατά πόσον είναι τα κατάλληλα οχήματα για ειλικρινείς ε, ανοιχτές συζητήσεις και ε, ελπίζουμε και λύσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε δράσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στις χώρες μας και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε συνεπώς και τι ε, ζωέ των πολιτών μας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουμε ε, πώς μπορούμε να άρουμε φραγμούς ε, στην αγορά εργασίας, να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, να μην υπάρχουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔ, να μπορέσουμε να έχουμε θέσει εργασίας για νέους ανθρώπους και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία από την οικονομία και τις επιχειρήσεις μας, ώστε η ευρωπαϊκή ε, οικονομία και να ανοίξει και να υπάρχουν ευκαιρίες για τους πολίτες. Έτσι ε, προωθούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το να συμβαδίζουμε είναι πάντα καλύτερο από το να βαθμολογούμε ο ένα τον άλλον. Δεν είμαστε αρχηγοί ο ένα του άλλου ή επικεφαλής ο ένα του άλλου, είμαστε εταίροι. Δεν χρειαζόμαστε νέους τρόπους για να απειλούμε ο ένα τον άλλον, χρειαζόμαστε τρόπου για καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη εφαρμογή και καλύτερους και θετικότερου να συνομιλούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόφι Ινεντβέλτε έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και τον Επίτροπο Τίμερμαντς. Είμαι λίγο απογοητευμένη πρέπει να πω, διότι ο κύριος Τίμερμαντς είπε ότι δεν χρειαζόμαστε ε, συνεχή θεσμική συζήτηση για τους μηχανισμούς. Εγώ θεωρώ ότι επακριβώς ε, αυτό χρειαζόμαστε, διότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις εξίες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται στο άρθρο 2 των συνθήκων. Είναι το πιο σημαντικό άρθρο. Είναι το σημαντικότερο ιεραρχικά άρθρο και ε, η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου από εκεί και πέρα μειώνεται από όλα τα άρθρα στη συνθήκη. Στη συζήτηση για την Ευρωζώνη είχαμε πει τότε ότι δεν χρειαζόμαστε δεσμευτικά μέσα στην Ευρωζώνη γιατί έχουμε συμφωνία κυρίων όλα τα κράτη-μέλη απλώ θα πρέπει να τηρήσουν τι δεσμεύσει του. Είδαμε σε τι μα οδήγησε αυτό και νομίζω ότι ήγηκε και η ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρχίζει να εξελίσσεται σε μία πολιτική ένεση, να ε, διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να εφαρμόσει αυτέ τι αξίε για τι οποίε είναι τόσο περήφανοι. Δεν θα πρέπει απλώ να μιλούμε, να μην είναι μόνο λόγια, ακόμα και αν είναι σε πέντε ή έξι γλώσσες, αγαπητέ Επίτροπε, θα πρέπει να υπάρχει δράση σε όλε τι γλώσσε και πραγματικά χρειαζόμαστε δεσμευτικά μέσα. Όχι απλώς συμβάσεις και σιωπηλή ε, διπλωματία και ε, συζητήσεις. Ε, χρειαζόμαστε μέσα. Γι' αυτό και η ομάδα μου, η Φιλελεύθερη, είναι το σύμφωνο της Δημοκρατικής Διακυβέρνησης. Το υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το συζητούμε έκτοτε θεωρούμε ότι μπορεί να εγκριθεί επί τη βάση των κείμενων συνθήκων και θα αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Είναι κάτι αντίστοιχο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε εφαρμογή των αξιών που μα ε, ε, χαρακτηρίζουν όλους. Και υπάρχει ένα μέσο, θα σας το δείξω, ε, είναι μια κάρτα, ένας πίνακας βαθμολόγησης και εκεί έχουμε βαθμολογήσει και τα 28 κράτη-μέλη με βάση κάποιους δείκτες. Για παράδειγμα, ελευθερία του λόγου, ελευθερία του συναθρίζεσαι, η μεταχείριση, ανεξιθρησκεία. Ε, και ήμασταν πολύ καλοί. Δεν έχουμε βάλει τα ονόματα των κρατών μελών. Απλώ να σα πω ότι αυτοί που είναι στο πράσινο είναι η Δανία και η Σουηδία και τα υπόλοιπα κράτη θα παραμείνουν ανώνυμα. Εάν γίνει αυτή η διαδικασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα Εθνικά Κοινοβούλια κάθε χρόνο και εδώ ε, δέχομαι και την πρότασή σας για μια ετήσια συζήτηση, η οποία θα γίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα θεσμικά όργανα για την κατάσταση της δημοκρατίας του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί εδώ ε, συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο, θα πρέπει να τη χάνουν ίσης μεταχείριση σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, μηχανισμοί ελέγχου για κάθε κράτος μέλος ή μόνο για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ή μόνο τα υποψήφια κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγχονται. Δεν θα ελέγχουμε μόνο τον προπολογισμό τους, δεν θα ελέγχουμε μόνο το χρέος και το έλλειμμα, αλλά θα ελέγχουμε και το κατά πόσον εφαρμόζονται οι κοινέ μας αξίες και θα κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινότητα των αξιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγο στον κύριο Χρυσόγονο για ένα λεπτό. Η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα οποία υποτίθεται ότι στηρίζεται η ευρωπαϊκή ένωση σύμφωνα με το άρθρο 2 της ιδρυτικής της συνθήκης αμφισβητούνται σήμερα στην πράξη από τα ίδια τα όργανα της ένωσης. όταν η ευρωπαϊκή επιτροπή απαντά γραπτώς σε ερώτησή μας ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν ισχύουν στα πλαίσια των μνημονίων αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες των κρατών μελών της ένωσης τα οποία τελούν υποκαθεστώς μνημονίου αντιμετωπίζονται ως ευρωπαίοι δεύτερης κατηγορίας και τα κράτη αυτά ως απικίες χρέους. όταν ακόμα ο επίτροπος κατάινεν δηλώνει ανερυθρίαστα ότι δεν αλλάζουμε πολιτική ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών αυτό υποδηλώνει περιφρόνηση για τη δημοκρατία. οι δικτάτορες του 20ου αιώνα παρεμπόδιζαν τη διενέργεια εκλογών με τη χρήση στρατιωτικής βίας ενώ ο μετανεωτερικός αυταρχισμός των ευρωπαϊκών ελίτ του 21ου αιώνα επιχειρεί ουσιαστικά να ακυρώσει τις εκλογές μέσω οικονομικού εκβιασμού. η ευρώπη χρειάζεται αλλαγή πορείας. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Προεδρία μας εξήγησε ότι το Συμβούλιο θα ήθελε να γίνεται μια φορά το χρόνο συζήτηση για την κατάσταση πραγμάτων της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Η κυρία Ζίπελ είπε ότι θα είναι ένα γεύμα. Και ο Επίτροπος Τίμεμανς μας είπε μόλις τώρα ότι δεν θέλει να έχει κομματική γραμμή για το θέμα αυτό. Δυστυχώς έκλεισε το μικρόφωνο. Συνεχίζει η κυρία Σαρτζεντίνη. Μας είπε ότι θέλει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος. Σαν διαιτητής σε αγώνα. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, ότι ο διαιτητής ε, έχει κανόνες βάσει των οποίων ασκεί τη δραστηριότητά του. Αλλά εμεί εδώ δεν έχουμε κανόνε ακόμη. Δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώ είναι αυτοί οι κανόνε Για το πώ θα εξετάζουμε ε, εάν υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν έχουμε κανόνε γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να διατυπωθούν. θα πρέπει επιτέλους να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να το τολμήσουμε αυτό. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε πραγματικά το πρόβλημα. Γιατί μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Παράλληλα, πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα ελευθερίας του τύπου, τα θέματα της ελευθερίας του συνέρχεστε και άλλες διακρίσεις. Και αυτό σίγουρα δεν συμβαίνει. Και αν δεν υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κανόνες, γιατί να θέλει κανείς να ενταχθεί σε ένα τέτοιο κλαμπ, σε μια τέτοια λέσχη. Διότι το θέμα είναι ότι πριν ενταχθεί, ε, υποτίθεται ότι πρέπει να συμμορφωθεί με κάποιε υποχρεώσει, αλλά άμα μπει μέσα, μετά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διότι δεν εφαρμόζονται οι ισχύοντε νόμοι, γιατί δεν υπάρχει στο Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο υπαρκή πολιτική βούληση. Και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και ελπίζω η Λετωνική Προεδρία να κάνει επιτέλου κάτι για το θέμα αυτό προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ η κυρία Φεράρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ της νομικής αναγνώρισης και της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρά τα άρθρα 2, 6 και 7 των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα δεκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Βλέπουμε τις αρνητικές και καταστροφικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της πολιτικής λιτότητας, παράνομων δραστηριοτήτων όπως η διαφθορά και διάφορες μορφές εγκληματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κατεπηγόντω μια εσωτερική στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου, ώστε να διασφαλίσει και συνέπεια με το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο προβλέπεται επί του ζητήματο στι εξωτερικέ σχέσει. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας μηχανισμός για να αξιολογήσουμε αποτελεσματικά τη μέρημνα και την προώθηση ε, των ε, κοινών ευρωπαϊκών αξιών που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή και στην εθνική νομοθεσία. Το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης έμεινε νεκρό γράμμα και ο εναλλακτικό μηχανισμός που προσφάτως μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη ανακοίνωση για το κράτος δικαίου δεν είναι καθόλου φιλόδοξο προκειμένου να ε, υπάρξει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προσβλέψουμε αποτελεσματικά διαφορετικές μορφές παρακολούθησης και ένα σύστημα κυρώσεων όταν διαπιστώνονται ότι υπάρχει παραβίαση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά έργανα και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα υποβάλλονται σε μια ε, στενα, ε, ε, διεξοδική ανάλυση ώστε να μην συνεισφέρει η Ευρώπη είτε έμεσα είτε άμεσα στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην επικράτειά της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέναρς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν αρκετά πράγματα ήδη, αλλά το κράτος δικαίου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μας ενώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι αυτό για το οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε. Και αυτό όχι μόνο για τους πολίτες μας, αλλά και για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Όταν αναφερόμαστε σε ε, άλλες χώρες, σε ανθρώπους με τους οποίους ε, συνάπτουμε συμφωνίες και εταιρικέ σχέσεις, πάντα αναφερόμαστε στο κράτος δικαίου. Αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει δημοκρατία και ούτε και η οικονομία δεν έχει αποτελέσματα. Επομένω, θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε. Θα πρέπει να μπορούμε να τηρούμε ε, τα του οίκου μας. Ε, και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, κύριε Τίμερμανς, διότι πριν από δύο χρόνια ήσασταν υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και αποστήλατε μία επιστολή επί του ζητήματο και συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να ασχοληθούμε με τι θεμελιώδει ελευθερίε. Πριν ένα χρόνο αργότερα, σα συνεχάρισαν στα πλαίσια των ε, συνθήκων για τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν οι συνθήκες και ξεκίνησε εργασία επί του ζητήματος. Αλλά το ερώτημά μου, κύριε Τίμερμανς, είναι το εξή. Αποστήλατε αυτή την επιστολή πριν από δύο χρόνια. Αν δείτε την εμπειρία σας, ιδιαίτερα ένα χρόνο μετά τη νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη δημοσίευσή σας, είστε ικανοποιημένος, είστε ικανοποιημένος με αυτά τα οποία έχουν γίνει. Υπάρχουν δυνατότητες στο παρόν πλαίσιο να γίνει κάτι περισσότερο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες ανεξάρτητα από το που βρίσκονται, τι κυβέρνηση ε, είναι στην εξουσία ε, μπορούν πραγματικά να έχουν ε, στις πρώτες προτεραιότητές τους τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος την Κιλάρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, πολλές φορές έχετε μιλήσει στο Κοινοβούλιο για να πείτε ότι αυτό που ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κρίση έγινε κοινωνική κρίση λόγω της ε, όξυνσης των ανισοτήτων και έγινε πολιτική και ηθική κρίση διότι υπάρχει απόγνωση και το συνέστημα της απόγνωσης που ήταν η βάση για να αναπτυχθούν οι ιδέες αυτές, οι αντιευρωπαϊκές της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Και αυτό σημαίνει πως η κατάσταση των ανθρωπίνων, ε, των, ε, του κράτους δικαίου είναι εν κινδύνο. Βεβαίως ε, η, ε, το βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Ένωσης είναι το άρθρο 2 που μιλάει για τις βασικές μας αξίες. Το κράτος δικαίου, η αξιοπρέπεια των ατόμων, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ο σεβασμός των μειονοτήτων. Αυτά είναι τα βασικά. Πρέπει λοιπόν σαφέστατα να τονίσουμε ότι το κράτος δικαίου και η ποιότητα της δημοκρατίας μειώνονται στην Ευρώπη γιατί δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να εγγυώνται την ουσιαστική εφαρμογή των αρχών αυτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το περίφημο δίλημα της Κομπεχάγης. Υπάρχουν ε, έλεγχοι όταν εντάσσεται μια χώρα, αλλά άπαξ και ενταχθεί δεν υπάρχει κανένα έλεγχο για το κατά πόσον διατηρούνται αυτέ οι προδιαγραφέ. Η προστασία των μειονοτήτων και η απαγόρευση των διακρίσεων και των διώξεων κατά των μειονοτήτων. Δεν αρκούν οι αρχέ ε, στην ανακοίνωση τη Κομισιόν του 2014 ούτε ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών μέσω του Συμβουλίου. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικού μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στην προσπάθεια πυθού και των διαδικασιών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7. Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο αυτή τη στιγμή να εφαρμοστεί το άρθρο αυτό. Πρέπει να βρούμε μια μέση οδό μεταξύ της προσπάθειας να πείσουμε μια χώρα και της ε, εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται στο κράτος στο άρθρο 7. Διότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ποτέ δεδομένη τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Σκρίπεκ. 1,5 λεπτό. Ευρωπαϊκή Aj na margo svojich predrečníkov o kontrole a dohľade tu prirodzeným priestorom pre rozvoj demokracie a ľudských práv sú... όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι κανείς ε, ε, δεν θέλει να αμφισβητεί τέτοιου είδους δικαιώματα. Οποτεδήποτε υπάρχουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συζητούνται. Φοβούμε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να εισάγουμε αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου απέναντι στα κράτη-μέλη. Γνωρίζω βέβαια ότι όπου σταματάει η συζήτηση ξεκινάει η δικτατορία των ε, επιταγών, των επιτακτικών εντολών. Γι' αυτό λοιπόν ε, περιμένω από τους συναδέλφους ευρωβουλευτές ανεκτικότητα και σεβασμό και ερωτώ έχουν όλοι όσοι ανήκουν στην οικογένεια τη δική μας την άποψη ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για τη δημοκρατία. Τα κράτη-μέλη έχουν τους μηχανισμούς για την προστασία της δημοκρατίας και αυτά πρέπει να γίνονται σεβατά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα περισσότερο σεβασμός και λιγότερο έλεγχος. Να υπάρχει τήρηση της και σεβασμός της ε, κυριαρχίας των κρατών μελών. Σεβασμός λοιπόν αντί για καταστολή. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτή η άποψη στο έγγραφό μας και να διαγραφεί το ενδεχόμενο της επιβολής κυρώσεων απέναντι στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μία μπλε κάρτα, ε, τη δέχεστε, παρακαλώ. Κύριε Βουλευτά, δεν με εξέπληξαν αυτά που είπατε. Πριν από λίγες ημέρες απευθυνθήκατε στους ευρωβουλευτές και στραφήκατε, είπατε ε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα απέναντι στη Σλοβακία για το δημοψήφισμα που διοργάνωσε. Μα πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά γίνονται για να προστευτούν προστατευτούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Πώς μπορούν λοιπόν αυτά να συμβαστούν με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διακριτική μεταχείριση έναντι των μειονοτήτων. Και πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, αυτό καθευτό, τι, ποιες είναι οι μειονότητες. Διακόπη δυστυχώς η απάντηση. Υπάρχει μια δεύτερη μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Ευχαριστώ. Είπατε ότι επιβάλλονται αξίες και δικτατορίες. Αλλά δεν ισχύει ότι το δημοψήφισμα αυτό απέτυχε. Και ευτυχώς θα λέγα γιατί μόνο 20% θεώρησαν ήταν αναγκαίο να ψηφίσουν. Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού στη Σλοβακία σέβονται πολύ περισσότερο τα άτομα των σεξουαλικών μειονοτήτων από ότι εσείς μοιάζει να θεωρείτε. Κυρία συνάδελφε, όποιος θέλει να πάει στην κάλπη, αυτό είναι θέμα των ε, ψηφοφόρων. Αλλά η καμπάνια που έγινε κατά του δημοψηφίσματος ήταν άδικη ήταν απαράδεκτη, ήταν μυσαλόδοξη. Και γι' αυτό πρέπει να καταγγείλω ότι υπέστη πίεση ένα κυρίαρχο κράτος. Αυτά είναι θέματα ηθικής, αυτά είναι θέματα οικογενειών και για κάθε κράτος πρέπει να υπάρχει κυριαρχία για τα θέματα αυτά. Και όσον αφορά το δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα αυτό είναι έκφραση ε, το, της Βούλης των Ψηφοφόρων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πολύ υψηλέ προδιαγραφές για την ε, λειτουργία της. Πρέπει να σέβεται κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, πρέπει να λειτουργεί το κράτο δικαίου. Αλλά όλα αυτά είναι προδιαγραφές που θέτει για την ένταξη στη χώρα. Αλλά όταν κανείς ενταχθεί στην Ένωση, μετά δεν υπάρχει καμία διαδικασία συνέχισης του κατά πόσον συμμορφούται η χώρα. Και αυτό είναι αυτό που αποκαλούμε το δίλημα της ε, Κοπεχάγης. Έχουμε μια σειρά από παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα χωρών όπου δεν υπάρχει ελευθερία ε, των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στη Λιθουανία δεν σέβονται την ελευθερία του τύπου και στη Ρουμανία υπάρχουν διακρίσεις κατά τον Ρωμά. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε να προτείνουμε κυρώσεις κατά χωρών που δεν σεβάστηκαν οικονομικές συμφωνίες. Αλλά όταν πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Επιπλέον, θα πρέπει να έρθει η στιγμή να τιμωρηθούν και οι χώρε που περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα και έχουμε και αυτό το πίνακα με τη βαθμολογία για το κατά πόσο τα πάνε καλά τα κράτη-μέλη στα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε τα λόγια μας πράξη. Δέχεστε μία μπλε κάρτα, κυρία Βουίξτρομ. Ευχαριστώ λέει η κυρία Βουίξτρομ. Ο κύριος Μπουντά. Το μικρόφωνο σας κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ρωτήσω την κυρία Οίλστρεμ, ξέρει ότι στη Ρουμανία όλες οι εθνικές μειονότητες έχουν τη δυνατότητα να έχουν σχολική εκπαίδευση στη γλώσσα τους. Και νομίζω ότι είναι υποδοματική από αυτή την άποψη για όλη την Ευρώπη η Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Βίξτραμ. Εάν η Ρουμανία, εάν ε, στη Ρουμανία υπάρχουν δυνατότητε εκπαίδευση σε όλε τι ε, γλώσσε, αυτό είναι θετικό. Αλλά ξέρω πόσο πολλοί ζητιάνοι Ρωμά ζητιανεύουν στην Ουψάλα. Μέτρησα 32 ε, ζητιάνου Ρωμά από τη Ρουμανία σε μερικέ εκατοντάδε μέτρων που ζη, ζητιάνευαν μέσα στην ε, χιονοθύελα και αυτό ε, είναι αποτέλεσμα των διακρίσεων που βρίσκονται στη χώρα σας. Ευχαριστώ η κυρία Λούνασεκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνάδελφοι. Ο κύριος Κρίπεκ είπε ορισμένα που με επίθυνε ότι πρέπει να μιλήσω για τις διακρίσεις κατά των ομοφιλοφίλων και των άλλων σεξουαλικών μενοτήτων και είπατε ότι φέστη πιέσει σε ένα κυρίαρχο κράτο η Σλοβακία. Αλλά κανεί δεν πίεσε την ε, Σλοβακία και το κοινοβούλιο τη να αποφασίσουν να οργανώσουν δημοψήφισμα κατά των δικαιωμάτων διενοτήτων. Αλλά δεν, και δεν ισχύει αυτό το οποίο ε, είπατε. Ε, η, δική σας προπαγάνδα αξιοποίησε ακόμη και τον Πάπα. Λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριο Τίμερμαν, χρειαζόμαστε ένα οδικό χάρτη για να κατονομήσουμε την ομοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε νόμους, αλλά δεν έχουμε διαδικασίες που να βοηθεί τους ανθρώπους των σεξουαλικών μειονοτήτων να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν έχουν αρκετή ενημέρωση. Η Λιθουανία απαγόρευσε ένα βιβλίο με παραμύθια που δείχνει ανθρώπους τέτοιου διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανισμούς επιτήρησης για να είμαστε σίγουροι ότι οι θρησκευτικέ μειονότητες ε, δεν υφίστανται διακρίσει. Κύριε Σκρίπεκ, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα διάλογο. Ο ομιλητής ο κύριος Σόγκορ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους ε, τα θέματα των, ε, ε του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ μιλάμε ανοιχτά, αλλά μέχρι τώρα εμπειρία έχει καταδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεφεύγει από αυτό το θέμα και λέει ότι δεν είναι αρμόδια. Και το Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών και δεν εξετάζει ποτέ τίποτα σε βάθο. Βεβαίω, και είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε σκληρά για την εμπιστοσύνη των πολιτών και γι' αυτό μιλάμε ανοιχτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για δημοκρατία και ευνομούμενα κράτη, τότε πρέπει να λέμε και για ποια κράτη μιλάμε που δεν εφαρμόζουν και δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν μιλάμε για ε, ευνομία ε, θα πρέπει να ακούμε και την άποψη των μειονοτήτων και να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις διαμαρτυρίες τους γιατί αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι η Ευρώπη ανήκει στους πολίτες της μόνο εφόσον δεν συγκαλύπτονται τα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τις εθνικές μηνότητες η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Ρουμανία βρίσκονται στην τελευταία θέση ως προς την προστασία των δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση για το κράτος δικαίου ε, μπορεί να τελεσφορήσει μόνο εφόσον η Κομισιόν και το Συμβούλιο εξετάσουν τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την γενική εικόνα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τους ε, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσον τον ειστερνίζονται ή όχι. Κάποια κρατημέλη δεν θα χαρούν για όλα αυτά. Αν όμως δεν διεξάγεται διάλογος, τότε κατ' ουσίαν η Ευρωπαϊκή Ένωση ομολογεί ότι δεν μπορεί να συμβάλλει στη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην επικράτειά της. Ο κύριο Τζαμπάσκη έχει μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, πρέπει η εσωτερική τάξη σε κάθε χώρα να ορίζεται από τη σύνθεση του λαού. Νομίζω ότι είναι ανταπαραγωγικό να προβαίνουμε σε παρεμβάσεις και γενικεύσεις. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Δύο λεπτά η κυρία Κόφμαν. Ε, η κυρία Κόφμαν. Χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου να γίνει πολιτικό διάλογο για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου και τη διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστούν παραβιάσει συστηματικέ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Και δύο είναι θετικέ εξελίξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μία κοινή αγορά, βασίζεται σε κοινέ αξίες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρά αποτελεσματικά για την προστασία αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Μόνο όποιος ε, έχει ρυθμίσει τα του οίκου του μπορεί αξιόπιστα να κατηγορεί τρίτους. Και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν εκπτώσεις. Εφόσον είμαστε κοινότητα αξιών πρέπει να σεβαστούμε και την αρχή της μη πρέπει να δεχθούμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε διότι τα κράτη μας είναι τόσο στενά συνδεδεμένα που οι εθνικές πολιτικές είναι τμήμα της ευρωπαϊκής εσωτερικής πολιτικής. Όμως αγαπητοί συνάδελφοι, τα μέτρα της Επιτροπής και του Συμβουλίου πάνε προς σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει να συμπληρώσω ότι είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Πραγματική προσπάθεια σεβασμού των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν υπάρχει ακόμη. Θα γίνεται μια φορά το χρόνο συζήτηση και από ό,τι φαίνεται και κλεισμένο των θυρών. Θα πρέπει λοιπόν ε, τα άλλα δύο θεσμικά όργανα να δουν τι προτάσει του Κοινοβουλίου ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό Κοπενχάγη. ένα δηλαδή μηχανισμό που θα επιτηρεί την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου τακτικά μέσω ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων και με βάση αντικειμενικά στοιχεία και δείκτες. Χρειαζόμαστε ουσιώδη ε, μηχανικό έλεγχο των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως κάνουμε στα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Μαούρα Μπαραντιάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση μας ε, ε, δημιουργεί την ανάγκη να κάνουμε αυτοκριτική. Αυτοκριτική γιατί συνεχίζουμε να μιλάμε για την προάσπιση της ελευθερίας έκφρασης ως μια αυθεντικά ευρωπαϊκή αξία και μπορούμε να πούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη τηρούν το άρθρο 11 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σας παραθέτω, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία τους. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το εθνικό τηλεοπτικό κανάλι είναι μέσω προπαγάνδας της κυβέρνησης Ορμπάν υπάρχει φόρος για τα έσοδα από τη διαφήμιση για να ελέγχονται τα ιδιωτικά μέσα επικοινωνίας και της αντιπολίτευσης και οι δημοσιογράφοι ε, πλήττονται από μια ε, ανήκουστη ε, πίεση. Και δεν το λέω εγώ, το λέει μια πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που επιβεβαιώνει ότι τα δημοκρατικά πρότυπα και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία βρίσκονται σε σαφή παναχώρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να παιδίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να διασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριο Γιάβορ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η συζήτηση για τα δικαιώματα αυτά δεν ε, έχουν ε, επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως ε, πρέπει να λάβει μέτρα όσον αφορά αυτή την κατάσταση στην Ουγγαρία. Αναφερθήκαμε στους μηχανισμούς ε, που είναι απαραίτητοι για να επιβάλλονται κυρώσεις. Θα ήθελα όμως ε, να υπογραμμίσω και κάτι άλλο. Όσο δεν έχουμε μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για το ότι σε μεμονωμένα κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο δεν υπάρχει αυτό δεν μπορούμε και να δίδουμε μια ουσιαστική απάντηση. Οι διαδικασίε, τα μέτρα, αν θέλετε, που έχουν ληφθεί σε σχέση με την Ουγγαρία έχουν επικριθεί επανειλημμένα. Όσο όμως ε, όλα αυτά είναι σε πολιτικό επίπεδο, οι συζητήσεις απλά εξαρτώνται από τις πολιτικές που ακολουθούνται. Ο κύριος ε, Πάμπεξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση δείχνει κατ' ουσίαν ότι δεν είμαστε τέλειοι θεσμοί, ούτε τέλειες κοινωνίες, αλλά ούτε και τέλειες χώρες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μερικές φορές ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι τα θεμέλια των θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε όμως την ιστορία μας θα δούμε ότι διαφορετικά εφαρμόζονται τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα στη Δύση, αλλιώς στην Ανατολή, αλλιώς στον Νότο. Δεν μιλάω τώρα για τον ε, ε, πρόδρομο των Ηνωμένων Εθνών, ε, ούτε μιλάω για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι η Σλοβακία. Το ίδιο ισχύει και για χώρες ε, οι οποίες προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης και τα οποία εφαρμόζουν και προστατεύουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Θέλω λοιπόν να πω το εξή, ότι θα πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι όχι μόνο στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και σε άλλε αρχέ που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Την αρχή του Μοντεσκιό, διάκριση των εξουσιών εφαρμογή του νόμου, τα δικαστήρια είναι στη τελική ανάλυση εκείνα που αποφασίζουν και όχι οι πολιτικοί θεσμοί. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συστήσουν πολιτικούς θεσμούς που θα αναλάβουν το ρόλο των δικαστηρίων, θα τα αντικαταστήσουν. Εγώ αυτό το βρίσκω αντιπαραγωγικό. Και ας μην ξεχνάμε ότι και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκείνου οι οποίοι επηρεάζονται από ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται και από κόμματα που χρηματοδοτούνται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές καθόλου δεν ενδιαφέρονται ούτε για θεμελιώδη δικαιώματα, ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για οτιδήποτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ ε, διαμαρτυρόμεθα. Γι' αυτό λοιπόν ας χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε, ας παραμείνουμε πιστοί στην διάκριση των εξουσιών και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει πολύ καλύτερα από ό,τι τα καταφέραμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Κινίτση για δύο λεπτά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τα ευρωπαϊκά συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων, αυτό το οποίο υπήρχε και αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο, αποτελούν ε, στοιχεία διαφύλαξης της δημοκρατίας και θέλουν να διασφαλίσουν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν ακόμα κενά και αδυναμίες στα συστήματα αυτά. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για παράδειγμα, εφαρμόζεται μεν στα κράτη-μέλη, αλλά μόνο στα πλαίσια του δικαίου της Ένωσης. Πρόκειται για μια ε, ε, συζητήσιμη ε, δυνατότητα τα περιορισμού που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε θέματα προ... Ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διαδικασία επιπαραβάσει, για παράδειγμα, από αποτελεί μέσο μόνο για συγκεκριμένες παραβιάσεις, ενώ επιτρέπει συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να απειλούν το κράτος δικαίου. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες του άρθρου 7 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιπτώσεις τις οποίες υπάρχει προφανής κίνδυνος ε, σοβαρής παραβίασης ή σοβαρής παραβίασης ε, κατ' επανάληψη των αρχών αυτών. Η ιδέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να ξεκινήσει το διάλογο για τα θεμελιώδη δικαιώματα εκτιμάται ιδιαίτερω και θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση σε κάθε περίπτωση συστημικής ε, παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ή αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το κράτο δικαίου και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει καλύτερα την έννοια του κράτου δικαίου και να το συνδέσει με κάποιε βασικέ αρχέ οι οποίε συνδέονται στενά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, σε γενικές γραμμές εκτιμούμε το συνολικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει όμως να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν, από, ξεκινώντας από περιπτώσεις οι οποίες ανησυχούν ιδιαίτερω, ε, για να μην υπάρχει διάκριση, περιθωριοποίηση και δίωξη και οποιαδήποτε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Παγκάθα Ουρτούντουα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα η διαφάνεια και η σωστή πρακτική στην δημοκρατική διακυβέρνηση θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και για να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η απαξίωση της ε, παραδοσιακής πολιτικής έχει να κάνει με αυτή την έλλειψη διαφάνειας και τις κακές πρακτικές. Σαν η πολιτική εμείς να είμαστε πάνω από τους πολίτες και όχι στην υπηρεσία τους. Ο μηχανισμός του άρθρου 7 δεν βασίζεται το άρθρο 2 των συνθήκων Ορισμένε από τι κακέ πρακτικέ έχουν να κάνουν με την πολιτικοποίηση ορισμένων εξουσιών που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητε. Και αυτό επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η πολιτικοποίηση των δικαστικών αρχών και του ελέγχου των ταμιευτηρίων μα κόστησε το διπλάσιο από όλε τι περσινέ περικοπές σε χρήμα αλλά και σε κοινωνικό έλεγχο. Η κακοδιακυβέρνηση μας κάνει πιο φτωχούς και λιγότερο ελεύθερους. Γι' αυτό κύριε Τίμεμανς πρέπει να κάνουμε μία παρατεταμένη και αναγκαία συζήτηση. Η κυρία Μακοβέ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε κράτος δικαίου. Οι πολίτες και οι κυβερνώντες πρέπει να σέβονται τον νόμο. Το κράτος δικαίου αφορά τη σχέση μεταξύ των ιδιωτών μεταξύ τους και όχι μόνο μεταξύ πολιτών και κυβερνώντων. Κατόπιν, πώς θα πρέπει να καταλήγουμε σε νόμους, πώς, ποια είναι τα δικαιώματα των υπόπτων εγκλημάτων, πώς συλλέγουμε τους φόρους. Όλα αυτά, πώς καθορίζουμε τους φόρους, όλα αυτά είναι θέματα κράτους δικαίου. Το θέμα λοιπόν είναι πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Οι νόμοι, αν είναι να υπάρχει κράτος δικαίου, πρέπει να ε, εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο. Να είναι ίση για όλου. Και αν δεν υπάρχει κράτο δικαίου, δεν λειτουργεί η κοινωνία, δεν λειτουργεί η δικαστική εξουσία, η δημοκρατία και ούτε καν η κοινωνία. Το κράτο δικαίου είναι διαφορά μεταξύ δημοκρατία και δικτατορία. Δεν μπορεί να θεωρηθούν κάποιε παραβιάσει του κράτου δικαίου δευτερεύουσε. Όλε οι παραβιάσει είναι παραβιάσει. Τελεία και παύλα και κράτος δικαίου σημαίνει επίσης ότι πρέπει όλοι να συμπεριφερόμεθα με βάση τον νόμο. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου αν κάποιοι πολιτικοί αλλάζουν πολύ συχνά τον νόμο επειδή δεν τους αρέσει κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτημα, δεν τους βολεύει, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό έχουμε νόμους. Ούτως ώστε οι πάντες και οι πολιτικοί να προσαρμόζονται στο σεβασμό του νόμου. Όμως οι πολιτικοί επειδή μπορούν να αλλάξουν τον νόμο δεν χρειάζεται να προσαρμόζονται όταν δεν τους βολεύει ο νόμος. Το κράτος δικαίου σημαίνει επίσης να υπάρχει σαφήνεια δικαίου, να είναι προβλέψιμη η εφαρμογή τους, να εφαρμόζονται ταχαίως, ούτως ώστε όλοι να ξέρουν τι πρέπει να περιμένουν. Τα κοινοβούλια ως πρώτο πρωταρχικό καθήκον έχουν να ψηφίζουν σαφείς και ευεφάρμοστους νόμους. Δύο λεπτά για τον κύριο Νίντερμιλλερ. Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίως είναι υπερήφανο για το ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται κατ' ουσίαν ε, για την ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτώ, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα όταν ε, υποβάλλουν υποψηφιότητα. Αλλά τι γίνεται με τα κράτη-μέλη τα οποία είναι μέλη και δεν σέβονται τα δικαιώματα. Είπατε προηγουμένω ότι δεν υπάρχει ανελεύθερη δημοκρατία. Εγώ λέω ότι η Ουγγρική κυβέρνηση τάσεται υπέρ της ανελεύθερης δημοκρατίας. Κατανοώ βέβαια ότι έχετε κουραστεί ε, σχετικά με το θέμα των Ουγγρικών μειονοτήτων, αλλά τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ούτε η Κομισιόν ούτε το Κοινοβούλιο ε, δεν προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τι θα πούμε στους ε, πολίτες που δεν θα απολάβουν νομικής προστασίας. Και εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ε, συγκαλύπτουν την ανελεύθερη δημοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις τι να πούμε στους πολίτες μας Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να είμαστε δειλοί. Πρέπει να μαχόμετα ε, για αυτά τα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκασμένη αν θέλετε να αγωνίζεται για τα δικαιώματα αυτά και το δικό μας των καθήκον είναι να ε, βρούμε αποτελεσματικούς ε, μηχανισμούς Πρέπει σε ολόκληρη την Ευρώπη να ε, βρίσκουμε διαδικασίες ελέγχου, να είμαστε θαραλέοι και να κάνουμε και αποφασιστικά βήματα. Να μην είμαστε δειλοί, να μην ε, κρυβόμαστε γιατί αυτό θα ήταν το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη η κυρία Μπιλμπάου Βαραντίκα. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη είναι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις κατά της ασφάλειάς μας περικόπτοντας ελευθερίες. Ε, γιατί μας κόστησε πολύ η απόκτησή τους και η χρήση τους μας βελτιώνει. Και οι τρομοκράτες αυτό θέλουν, να τις καταργήσουμε. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερες δυνατότητες, ώστε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να εγγυώνται ότι όλα τα κράτη-μέλη θα σέβονται πάντα τις αρχές Κοπεχάγης. Συγχαίρω την Άλντε και ιδιαίτερα την αρμόδιά μας για τα θέματα ελευθεριών που υποστήριξε αυτές τις ιδέες στην πρόταση ενός συμφώνου για την δημοκρατική διακυβέρνηση και για την τρομοκρατία. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, θέλουν να υπάρχει η, η ποινή της, ε, των ισοβίων αναθεωρουμένων για ορισμένες ε, πολιτικές δραστηριότητες. Θα ήθελα να θυμηθούμε, όπως κάναμε σήμερα ε, για άλλες περιπτώσεις, να τονίσουμε ότι δεν έχει σεβαστεί η Ισπανία βασικές αρχές για την ποινική δικαιοσύνη. Η Ευρώπη χρειάζεται εργαλεία για να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε αποφάσεις δεν σέβονται την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κύριε Τίμερμαντ, πρέπει να δράσετε κατά των αποφάσεων της ισπανικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Βάιντενχόλτσα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Οικονομική Ένωση, είναι κυρίως Ένωση Αξιών. Και νομίζω αυτό αναφέρεται και στα κριτήρια της Κοπενχάγης το 1993. Έκτοτε όμως γίνονται πολλές συζητήσεις κατά πόσον τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε αυτά. Αυτό δημιουργεί πολιτικές διαφωνίες ε, και υπάρχουν φυσικά κάποιοι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων. Ε, η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική γιατί υπάρχουν μεμονωμένα κράτη μελη όπως στην περίπτωση της Ουγγαρίας, η οποία Ουγγαρία επιτρέπει στον εαυτό της να αγνοεί τις υποχρώσεις της. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως ένα μηχανισμό, ο οποίος ε, θα ε, επιβάλλει κυρώσεις. Δεν είναι σωστό να το αναβάλουμε αυτό διαρκώς. Κάτι τέτοιο θα ήταν και ζημιογόνο για την εύρυθμη λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ η κυρία Ρεβόντα Λόν Μπομφά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται σε αθεμελιώδεις αξίες οι οποίες είναι κοινέ ε, και ε, απαρέγκλητες. Η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτο μέλο πρέπει να πληρεί τα κριτήρια τη Κοπενχάγη για να διασφαλίζεται ο σεβασμό, η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτά τα κριτήρια δεν ισχύουν μόνο τη στιγμή τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να ισχύουν καθημερινά. Όμως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κρατημέλη. μελη Τα δικαιώματα και ελευθερίες πολλών ε, πολιτών παραβιάζονται, αγνοούνται ακόμα και στο ε, ε, εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωμά, η κοινότητα των ΛΟΑΔ, οι δημοσιογράφοι, ακόμα και οι μειονότητες και οι ετούντε άσυλο είναι άτομα τα οποία την χάνουν διάκριση, περιθωριοποίηση και κακομεταχείριση. Προκειμένου να επιβιώσει το πνεύμα της Κοπενχάγης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ε, να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο έλεγχος ε, θα πρέπει να γίνεται σε μια, ένα πλαίσιο συνεχούς διαλόγου για τα θεμελιώδη δικαιώματα και να υπάρχουν και ένα σύστημα κυρώσεων και ποινών πιο αποτελεσματικό η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 της συνθήκης που επιτρέπει να ε, μην υπάρχει δικαίωμα ψήφου ε, από ένα κράτος μέλος σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι μια κύρωση που πολύ δύσκολα μπορούμε να εφαρμόσουμε σήμερα. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα για να γίνονται σεβαστά τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Κυρία Μπομφά, υπάρχει μια μπλε κάρτα. Δέχεστε? Ο κύριος Ζεντόφσκι. Παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη μου έκπληξη άκουσα αυτά τα οποία ελέγχθησαν και πρέπει να σας πω, εγώ έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα ποδοπατούνται. Αν ισχύουν βέβαια όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Και αυτό ισχύει κυρίως για την κριτική που ασκήθηκε έναντι της Ουγγαρίας. Εγώ διαφωνώ ε, στεναρά και θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδεικνύουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην παράδοση, στη δημοκρατική παράδοση της Ουγγαρίας και τελικά εσείς τι, τι απαιτείτε, τι είδου μέτρα πρέπει να ληφθούν αυτό δεν ήταν μπλε κάρτα, αυτό κατ' ήταν ερώτηση θέλω να πω λέει η Πρόεδρος θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ Όσο υπάρχουν παραβιάσει των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί θα δίνουμε τη μάχη για να γίνουν σεβαστά. Και γι' αυτό θεωρούμε πω είναι απαραίτητο επιτέλου να έχουμε και το κράτο δικαίου στην Ευρώπη. Ο κύριο Κύρκο, είναι ο επόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πριν από λίγε μέρε ήμουν στην Τουρκία στα πλαίσια τη Μικτής κοινοβουλευτική επιτροπή, και εκεί προσπαθούσα να εξηγήσω στου Τούρκου συναδέρφου μου το σεβασμό του κράτου δικαίου αποτελεί προπόθεση για την προσχώρηση ενό κράτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία από τις κύριες αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση μαζί με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μου επισήμαναν όμω κάτι που και εγώ ήξερα. Υπάρχουν περιπτώσει που μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση του κράτου δικαίου δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και έτσι δημιουργείται απειλή για τη λειτουργία ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση ω χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Πώ λοιπόν ζητάμε από αυτού συμμόρφωση. Είναι αλήθεια πω τέτοιε περιπτώσει υπάρχουν πιστεύω λοιπόν ακράδαντα πω είναι απαραίτητο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο α πούμε μηχανισμό κοπενχάγη όπω αναφέρθηκε νωρίτερα που θα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με αντοχή στι πιέσει τέτοιε περιπτώσει μια και ο σεβασμό του κράτου δικαίου συνδέεται άρρηκτα με τη δημοκρατία. ευχαριστώ. Θα κάνουμε τώρα την διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 14 ε, βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Νομίζω 8 θα μπορέσουν να το κάνουν. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Σουνή. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα πρέπει να έχει σταθερού δεσμού και δημοκρατικό καθεστώ και κράτο δικαίου. Θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασία των μειονοτήτων. Αυτό περιλαμβάνεται στα κριτήρια τη Κοπενχάγη και η Σλοβενία έπρεπε να εκπληρώσει αυτά τα κριτήρια. Δυστυχώ, στη χώρα μου τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έχουμε την 24η επέτειο της ανεξαρτησίας μας, αλλά αντιμετωπίζουμε ακόμα προβλήματα μετάβασης. Και είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η σλοβενική δικαιοσύνη, η οποία έχει επιλεκτικό χαρακτήρα. Ορισμένοι μπορεί να καταδικάζονται επί τη βάση μονάχα ενδείξεων και άλλοι επί τη βάση στοιχείων τα οποία είναι ανεπαρκή. Και υπάρχει και το πρόβλημα ε, ποιότητος και ενότητος των δικαστικών αποφάσεων. Το δικαστικό σύστημα στη Σλοβενία αυτή τη στιγμή αποτελεί το κύριο εμπόδιο για μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. <clears throat> Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσει την κατάσταση της Σλοβενίας. Το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σηματοδοτεί μια τροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει πολλά, αλλά πολλά μπορούν, πρέπει να γίνουν ακόμα. Ο ρόλο που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, ε, δικαιωμάτων κατά οποιασδήποτε διάκριση για τα δικαιώματα των ε, γυναικών για την ισότητα των φύλων. Γι' αυτό ακριβώ χαιρετίζω ε, την παρέμβαση του Αντιπροέδρου Τίμερ μας. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε τελικά νομικά δεσμευτική. Η δράση της Ένωσης δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην απλή κύρωση. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό ε, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χώρο προστασία, προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση τον ορισμό ε, και τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα χώρο που δεν θα πρέπει να έχει ω όρια την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριο Μαρία, Ένα λεπτό. I will speak in Greek. Κυρία Τίτεμανς, η διγλωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ένωση είναι καταφανής. πριν λίγες μέρες στις 26 Ιανουαρίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών έθεσα το ζήτημα ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και ζήτησα από την Επιτροπή να αναλάβει δράση η οποία όμως δήλωσε αναρμοδιότητα καθώς το μνημόνιο δεν εμπίπτει δήθεν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση αυτή είναι πολιτικά και νομικά απαράδεκτη πολιτικά διότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ειδική ζώνη όπου δεν ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομικά διότι το μνημόνιο έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης με την απόφαση 2010 χιλιάδες του ecofin και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης στις 6 ιουνίου του 2010 στη σελίδα 9. θα συνεχίσετε λοιπόν τους ισχυρισμούς ότι μπορεί η τρόικα και το μνημόνιο να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ελλάδα; Ευχαριστώ. Članak Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι στο άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι κάθε μορφή μυσαλλοδοξία και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να κολλάζεται, ακόμα και στι περιπτώσει όπου αυτό γίνεται από κρατικέ αρχέ κάθε φορά που παραδιάζονται οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ενιαίος χώρος σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να αναστρέψω ορισμένα επιχειρήματα. Θα πρέπει να ασχίσουμε να μιλάμε για το να δίνουμε καλά παραδείγματα. Γιατί η Ευρώπη έχει πολύ θετικά παραδείγματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το γεγονός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θέλω να προτείνω να έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία, να εξάρουμε τα θετικά παραδείγματα και να τα κάνουμε γνωστά και στους εκλογείς μας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Εμείς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ηθική και πολιτική αυθεντία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κρίνει, λέει ο κύριος Βέγας, τη δημοκρατία σε οποιοδήποτε κυρίαρχο κράτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνει χώρες όπως η Κούβα και η Βενεζουέλα και υποτίθεται ότι υποστηρίζει μη κυβερνητικέ οργανώσει στι χώρε αυτέ, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτικέ φτωχοποίησεις και οδηγεί σε συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση της, του πλούτου στο έδαφο τη. Α είμαστε σαφεί λοιπόν. Βάσει τη τωρινή αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα είναι δημοκρατική μονάχα όταν κύπτει τον αφιένα ενώπιον των αγορών και των μεγάλων οικονομικών ομίλων. Αυτή είναι η πραγματική ε, κρίση. Αυτό είναι το πραγματικό κριτήριο που γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν οι λαοί να μπορέσουν να αποφασίσουν το μέλλον τους αυτόνομα χωρίς γεωστατικές, γεωστατικές ή οικονομικές θεωρήσεις που τους επιβάλλονται. Ο κύριος Μπάτεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται τώρα ανάγκη ενό πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και της ανθρώπινης δικαιοσύνη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε μια δημοκρατία ήδη από το 18ο αιώνα. Τώρα έχει γίνει κενό κέλυφο, γιατί οι περισσότεροι νόμοι μα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από το εκλεγμένο μα κοινοβούλιο. Έχουμε κράτο δικαίου, το οποίο έρχεται από την εποχή της Μαγνα Κάρτα, αλλά έχει ξεπεραστεί το αγγλικό ε, δίκαιο, το οποίο τώρα δεν υποχρε... αναγκάζονται να το αφήνουν να υπόκειται στην ε, υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου η... τα δικαστήριά μας. Μέτρα όπως το habeas corpus έχουν παρακαμφθεί από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Έχουμε δικαιώματα τα οποία με το σύστημα του κοινού δικαίου του Common Law έχουν εφαρμοστεί <clears throat> στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να μας διδάξει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος δικαίου και τα βασικά δικαιώματα. Η κυρία Γκάλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Με βάση τη δικαιοδοσία που έχουν. Το κράτος δικαίου μπορεί να υπάρξει και να είναι αποτελεσματικό αν αναλύει τα προβλήματα και ε, όχι όταν τα γεννάει τεχνητά. Προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά και όχι απλές καταγγελίες στο ΜΜΕ ή χαλκευμένες κατηγορίες. Έχουμε ακούσει να επαναλαμβάνονται και νέες ε, διακήρυξεις. Ε, δεν είναι η Ουγγαρία η οποία είναι ο κίνδυνος και δεν χρειάζεται να υπερασπίσετε τους Ουγγρούς πολίτες από την κυβέρνησή τους. Το καταλαβαίνουν όλα αυτά οι Ουγγροί πολίτες. Εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε σε πραγματικά προβλήματα, όχι ε, φανταστικά. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, Επίτροπε, ότι θα πρέπει να μας κρίνετε επίσης βάσεις. Και επίσης οι εθνικές μειονότητες θα πρέπει να προστατεύονται και να θεωρούνται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες. Ο τελευταίος ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε. Ήμουν κατ' επανάληψη σκιώδης εισηγητής για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ακριβώς με αυτή την ιδιότητα μπορώ να κρίνω το επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζω ότι σε κάποιους τομείς είναι αρκετά αδύναμος αυτός ο, και υπαρκεί αυτός ο σεβασμός. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει σε τρίτες χώρες ότι δεν τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλει να τις τιμωρήσει, εάν το κάνουμε αυτό θα πρέπει και εμείς να έχουμε ένα σύστημα για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δημοψήφισμα στη Σλοβακία έχει αναφερθεί κατά επανάληψη εδώ. Εγώ είμαι περήφανη για τη Σλοβακία, γιατί μόνο το 20% των ε, πολιτών. Συγγνώμη, μόνο το 20% των πολιτών ε, εμφανίστηκε σε εκλογές. Αυτό δεν είναι καλό. Έχουμε ακούσει πολλές ε, διακηρύξεις, ε, έμπλες μίσους στη Σλοβακία. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Στα πλαίσια του ΚΑΤΣΙΑΙ, τελείωσε μάλλον το ΚΑΤΣΙΑΙ και τώρα ο Επίτροπος. Um, first of all, the um,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 Absolutely. You are knocking open doors, sir. At least as far as it Όσο λοιπόν σας αφορά, πρέπει να σας πω πως αυτό που άκουσα από τους ανεξάρτητους Έλληνες ήταν αντίστοιχα τέτοια σχόλια. Οπότε δεν θα ήθελα αυτό να το ε, άρο. Πάντω, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση με το κράτο δικαίου, θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε στι ανάγκε μα. Και αν υπάρχει πρόβλημα με το μηχανισμό, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κριθεί ω ανεξάρτητο μηχανισμό, έτσι ώστε να δούμε αν τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο πρόβλημα. Να δούμε δηλαδή υπάρχει ανεξαρτησία σε επίπεδο ε, δικαστικού σώματος ή με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εγώ είμαι με το μέρο σας, είμαι απόλυτα στρατευμένος υπέρ αυτού του θέματος, αλλά θα ήθελα να με βοηθήσετε οι μηχανισμοί που έχουμε να γίνουν αποτελεσματικοί, να τους δώσουμε μια ευκαιρία πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το κατά πόσο χρειαζόμαστε καινούριου μηχανισμούς. Επόμενος ο μιλητής είναι η εκπρόσωπος του Συμβουλίου, η κυρία Καλνίνα Λουκασέβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Έχω ακούσει τις απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Όπως είπα και στην αρχή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται όχι μόνο στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά βασίζεται και στο κράτος δικαίου. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η εσωτερική του ένωμη τάξη σέβεται τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πολιτικός διάλογος, ο οποίος έχει θεσπιστεί τον Δεκέμβριο του 2014, μέσα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων περιλαμβάνει το σεβασμό για το κράτος δικαίου και τόνισε και πάλι τη δέσμευση των κρατών μελών να διαφυλάξουν τα βασικά όπλα της δημοκρατίας. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι ο νέος διάλογος θα πρέπει να εξασφαλίσει την τήρηση της αρχής του ε, κράτους δικαίου και ότι θα παραμείνει αυτό κοινό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε πρόσφατα το θέμα της προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην <clears throat> Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η, απόφαση όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου 2014 έχει δημιουργήσει κάποιες αμφιβολίες για το θέμα αυτό. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε για τα ζητήματα αυτά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις μας. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την υποχρέωση να γίνει μέλος της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και όχι αυτό να είναι προαιρετικό. <clears throat> Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν και νέοι μηχανισμοί παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Και αυτό να γίνει στην πόλη μας εδώ το Στρασβούργο όπου βρισκόμαστε. Συμφωνώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά τη δυνατότητα που μας δίνουν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα και ο μηχανισμός που είναι ενισχύ. Έχουμε λοιπόν τα απαραίτητα εργαλεία, χρειάζεται απλώς να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι ο πολιτικός διάλογος έχει δυνατότητες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, συμμόρφωση με τις αρχές που διατυπώθηκαν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2014. Με τον τρόπο αυτό έχουμε η αξία <clears throat> και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι όπως είπε ο κύριος Τίμερ μας θα μπορέσει το δικαστήριο να μας δώσει νέες ιδέες και η Κομισιόν να τις ε, εφαρμόσει. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση.